και τα συμπεράσματα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κρίση δίνω τον λόγο για τέσσερα λεπτά στον κύριο Γκέρονς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πρώτα κρούσματα του έμπολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν πανικό στην κοινή γνώμη. Από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο όταν χιλιάδες άτομα που είχαν μολυνθεί από τον ιό του έμπολα ε, κατέληγαν σε θάνατο στην Σιέρα Λεόνε, στη Λιβερία και σε άλλε χώρε τη Αφρική. Η κρίση ε, απέκτησε συστημικό χαρακτήρα, καταρχήν διότι υπήρχε έλλειψη ε, σε ε, ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία αναγνώρισε την ύπαρξη ελλημάτων στην βραδύτητα αντίδρασή τη. Τρει χώρε κυρίω επλήγησαν από την κρίση και τονίζουμε τον ιδιαίτερα οξύ χαρακτήρα τη κρίση. Στις χώρες αυτές το 80% ζει σε ε, φτώχεια. Ε, μόλις τέσσερα χρόνια είναι ο χρόνος σχολικής ε, εκπαίδευσης των παιδιών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των 29 φορέων, δηλαδή της Επιτροπής και των 28 κρατών μελών. Ο διορισμός ε, του Επιτρόπου ε, Στυλιανίδη ως συντονιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση του έμπολα επέτρεψε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα και να βρεθούν λύσεις ε, και να δοθεί βοήθεια στις τρεις αυτές χώρες της Αφρικής, Λιβερία, Σιέρα Λεώνα και Γουινέα. Κάποια συμπεράσματα μπορούν ήδη να εξαχθούν από την κρίση. Ήδη οι ανθρωπιστικές οργανώσεις φάνηκε ότι έδρασαν ταχύτατα, ιδίως ε, οι γιατροί χωρίς σύνορα και ε, ο Ερθρός Σταυρός προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν τον πληθυσμό και ε, χαίρουν εκτίμηση από όλου. Η καταπολέμηση του έμπολα κόστησε τη ζωή 500 περίπου ε, ατόμων ε, που παρήχαν ε, υπηρεσίες υγείας για την καταπολέμηση του, του έμπολα. Αρκετά γρήγορα βρέθηκαν και κάποιες λύσεις όσον αφορά και τον εμβολιασμό. Ακόμη πρέπει να δούμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα συστήματα υγείας στις χώρες, στις συναπτυσσόμενες χώρες, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα συστήματα αυτά στην τύχη τους χρειάζονται βελτίωση. Θα πρέπει επίσης ε, να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος για την έρευνα και για την ε, ανάπτυξη όσον αφορά την καταπολέμηση των σπανίων ασθενειών βλέποντας ε, την τύχη που περιμένει τις, τους κατοίκους στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία για μια νέα έκθεση ε, σε στενή συνεργασία με τον συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριο ε, Στυλιανίδη, και παράλληλα θα χρησιμοποιήσουμε και την αποστολή που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αφρική στις αρχές Νοεμβρίου όχι μόνο τα συστήματα υγείας ε, αλλά και την οικονομία των χωρών αυτών θα πρέπει να φροντίσουμε διότι είδαμε ότι ε, κατέρευσαν οι οικονομίες ήδη από τις αρχές ε, της επιδημίας αυτής. τουλάχιστον 20% της εξωτερικής ε, επίσημης βοηθείας έχουμε ε, υποσχεθεί ότι θα την εφαρμόσουμε στην ανάπτυξη, ανάπτυξη κυρίως υποδομών, κυρίως ε, ανάπτυξη συστημάτων υγείας και υποδομών στα συστήματα υγείας. Ο ιός αυτός μπορεί να είναι, ένα έξυπνος, να είναι ένας έξυπνος ιός, ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί υπό διαφορετικές μορφές. Δεν πρέπει λοιπόν να εφησυχάσουμε. θα πρέπει η πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη να είναι μια διαρκής ε, αρχή, η οποία θα εφαρμόζεται ε, συνεχώς. Και δεν θα πρέπει ε, να ξεχνούμε να το ρόλο που πρέπει να παίξει η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιώργης. Ακολουθεί για την Κομισιόν ο κύριος Στυλιανίδης Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έντιμα μέλη. η Κομισιόν χαιρετίζει ε, ιδιαίτερα την έκθεση αυτή του κύριου Γκέρνς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρνς για το σημαντικό του έργο και ιδίως για την ε, αφοσίωση που έχει δείξει στον αγώνα κατά του έμπολα. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε ένα θαυμάσιο επίπεδο συνεργασίας και είμαι ιδιαίτερα ε, ευγνώμων προς τον κύριο Γκέρνς για αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέχει μια, για την, μια, έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη μάλλον όταν πρόκειται για την προώθηση και την υποστήριξη της οικουμενικής κάλυψης σε υγειονομικό επίπεδο. Πρέπει να στις χώρες να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη και να εξασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα των συστημάτων αυτών, ώστε να μπορούν να ελέγχονται οι επιδημίες, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η επόμενη τέτοια επιδημία. Η έκθεση αυτή παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η επιδημία της έμπολα. Έχουμε ακόμα δυστυχώς κάποιες ε, περιπτώσεις στην Γουινέα τις τελευταίες εβδομάδες. Θα πρέπει να παραμείνουμε επάγρυπνοι μέχρι ό,τι μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα βαθμό μηδενικό κρουσμάτων και να βοηθήσουμε τις χώρες οι οποίες έχουν επηρεαστεί να ανακάμψουν πλήρως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν υποσχεθεί πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό 900 2 δισεκατομμύρια, συγγνώμη. 900 εκατομμύρια από αυτά τα ποσά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ε, επιδημίας και την έρευνα. Επίσης, μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να αντιλήσουμε τα σωστά συμπεράσματα από την κρίση της ΕΜΠΟΛΑ. Η συνδιάσκεψη του Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, όπου ήταν παρόν ο κύριος Ανδρουϊκάητης και εγώ, κατέληξε σε σημαντικές συστάσεις. που θα βοηθήσουν και το Συμβούλιο για τα θέματα υγείας το Δεκέμβριο. Επίσης, ως συντονιστής για τα θέματα αυτά, θα τονίσω ποια είναι τα συμπεράσματά μας και θα παρουσιάσω ενώπιον του Συμβουλίου στο τέλος του χρόνου. Θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουμε στη συζήτηση των G7 για την έμπολα, όπως το έχουμε πράξει ήδη και ε, πρόσφατα με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Άντριου Κάιτης. Χαιρόμαστε ότι η δήλωση των G7 εκφράζει την ε, προσήλωσή μας στο να υπάρξει ένα ενισχυμένο υγειονομικό σύστημα το οποίο θα παρέχει τις βασικές υπηρεσίες και την ε, παροχή καθαρού ύδατος ώστε να μπορέσουμε εν καιρό να επιτύχουμε την πλήρη κάλυψη. Ευχαριστώ πολύ. όπως το έχει η έκθεση Το καθαρό πόσιμο νερό και η φροντίδα υγείας για όλους είναι απαραίτητα. Και συμφωνούμε όλοι δύο πάνω στο ότι η κατασκευή και η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων υγείας είναι απαραίτητη, είναι αδύρυτη ανάγκη για να γίνεται σωστή εποπτεία αλλά και περιορισμός οποιασδήποτε τέτοιου είδους κρίσης. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση από την κρίση αυτή. Πολλά θα μπορούσε κανείς ε, να ε, γράψει για την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε γρήγορη και ουσιαστική χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του ιού έμπολα, για έρευνα, για ε, ανάρρωση, για ανάκαμψη των συστημάτων υγείας, για αναδιοργάνωση των ε, συστημάτων οδικών και άλλων μεταφορών ε, στην Αφρική, αλλά και για να αποκοπούν οι διάδρομοι μετάδοσης. Έχουμε απασχολήσει πολύ σημαντικούς επιδημολόγους και έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο το EU MedVac System, αυτό το σύστημα το οποίο εφαρμόσαμε για όλους τους επαγγελματίες της υγείας. Ναι. Και σίγουρα υπάρχουν διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε ε, για τα πράγματα που δεν πήγαν και όχι τόσο καλά, ε, όπως καλά πήγε όμως η αεροδιακομιδή, MedVac. Σε γενικές γραμμές η διεθνής κοινότητα δεν είναι καλά προετοιμασμένη για μια παγκόσμια επίγουσα κατάσταση στον τομέα της υγείας και θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους τομείς. Να έχουμε στήριξη περισσότερη στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, να υπάρξει μεταρρύθμιση του οργανισμού αυτού και να ε, αναθεωρήσουμε τους διεθνούς διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν στον τομέα της υγείας. Και πιστεύουμε ότι η βοήθειά μας μπορεί να είναι καθοριστική. Δύσκολα είχα, με δυσκολία ε, στείλαμε γρήγορες και ταχείες ομάδες ιατρικής αντίδρασης. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό ιατρικό σώμα ε, σε, χρησιμοποιώντας τον εθελούσιο μηχανισμό των κρατών μελών τα συστήματα υγείας ε, στις, ε, ε, στους εταίρους μας είναι αρκετά προβληματικά και εμείς Θέλουμε να τα ενισχύσουμε. Σε κάθε περίπτωση ο ιός έμπολα διδάσκει ότι ε, δεν λειτουργήσαμε αρκετά περιεκτικά, αρκετά συλλογικά. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έχουν περισσότερες δυνατότητες οι χώρες, ε, η κάθε μία, κάθε αυτή. Πρέπει να έχουμε φροντίδα υγείας για όλους, αλλά και για τον έλεγχο της επιδημίας κάθε φορά που ξεσπάει ε, μια τέτοια πλειάδα κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλη υποχρηματοδότηση του τομέα της της και οι εγχώροι πόροι δεν αρκούν για να καλύψουν τα κενά. Πρέπει να είμαστε σωστά προετοιμα... προετοιμασμένοι και να καλύψουμε τις ιατρικές ανάγκες και γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, μια δημόσια χρηματοδότηση της υγείας έστω και κατελάχιστον 40 ε, χώρες ε, εξοδεύουν λιγότερο από 30 δολάρια αμερικανικά ανακεφαλή ανά έτος και είναι αληθινός αριθμός αυτός, πραγματικό νούμερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προγραμματίσει τη βοήθεια που δίδει ε, στον τομέα της υγείας χωρίς να αφήσει κανέναν στο περιθώριο. Να αντισταθούμε στις τάσεις, να αποσυρθούμε συλλογικά από τον τομέα της υγείας. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις χώρες που έχουν που είναι κάτω από το κατόφλι, το ελάχιστο κατόφλι κρατικής χρηματοδότησης. Πρέπει να έρθουμε να καλύψουμε αυτό το κενό και να λειτουργήσουμε με πιο προβλέψιμο τρόπο. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στηρίξουν μια παγκόσμια συντονισμένη ερευνητική, ε, παγκόσμια συντονισμένη ερευνητική προσπάθεια η οποία θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες και θα ασχοληθεί με τα κοινά στην έρευνα έναντι μελλοντικών επιδημιών. Η έρευνα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και μπορεί να ενισχύσει τα τοπικά συστήματα υγείας. Στηρίζουμε την παγκόσμια ερευνητική συνεργασία για τις λοιμώδεις νόσους, για την ετοιμότητα για αυτές, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για το συντονισμό ε, των ε, δωρητών και των χρηματοδοτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας ο κύριος Χωράης Αμπάουντς. Για ένα λεπτό. Ακριβώ όπω και με του πρόσφυγε η ανταπόκριση ευρωπαϊκή για το εμπολέ κατά τη γνώμη μου ήταν κάτι που έγινε καθυστερημένα και έγινε με άστοχο τρόπο γιατί κάποιε λίγε χώρε να αυτές παντέρασαν σωστά αλλά η εντέλεση των ε, υπολείπων λοιπόν, ήταν θλιβερή συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λόγο ούτω ώστε να είναι περήφανη για αυτό που έκανε και γι' αυτό τα μαθήματα που θα πρέπει να εξαγάγουμε μετά από κάποια <clears throat> τίμια ειλικρινή ανάλυση είναι ότι του πρώτου μήνε που ε, ακολούθησαν κατόπιν του συναγερμού από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Ε, υπήρχε κάποια παθητική στάση και αυτό εξηγεί γιατί είχαμε τόσο μεγάλη διάσταση σε αυτή την ε, επιδημία και γιατί ήταν έξω από κάθε έλεγχο η εξάπλωση. Και αυτό μας έδειξε πόσο αργό και ανεποτελεσματικό είναι το σύστημα της υγείας και ε, ο μηχανισμό μα για να αντιδράσουμε σε τέτοιε κατευθύνσει. Αλλά χρειάζεται να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε με εμβόλια και με ε, θεραπείες, αγωγές. Οπότε χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα βοήθειας και ε, αντίδραση στους κοινούς Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, παρακαλώ. Να μην χρησιμοποιείτε για ερωτήσει ε, την μπλε κάρτα γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ. Οπότε, ο κύριος Πόγκα για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σάχλα Γκέρενς για τη συνεργασία του κατά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης η οποία είναι σημαντική και η οποία κάνει τον απολογισμό της μεγάλης υγειονομικής κρίσης που έπληξε τη Δυτική Αφρική το Μάρτιο του 2014 με περισσότερους από 11.000 θανάτους. Η κρίση του ιού έπολα ανέδειξε τις αδυναμίες των αναπτυσσόμενων χωρών στον τομέα της υγείας. Είναι απαραίτητο οι Ευρωπαίοι, όλοι οι παράγοντες που είναι ενεργοί στο θέμα της αναπτυξιακή βοήθειας να ενισχύσουν τη βοήθεια που τελικά δίδουν στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε αυτές να ε, δημιουργήσουν ε, ε, επαρκή και αποδοτικά συστήματα υγείας και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο κατάρτισης ιατρικού προσωπικού και στους άλλους τομείς. Θα πρέπει το ιατρικό προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται στις κρίσεις που μπορεί να ξεσπάσουν. Κάτι που μου φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό είναι η ανάγκη να ενισχυθεί η διακυβέρνηση των αναπτυσσόμενων χωρών. Όσο πιο ανοργάνωτη είναι μια χώρα, τόσο λιγότερο δυνατό είναι να έρθει κανείς να βοηθήσει τα θύματα. Χωρίς χρηστή διακυβέρνηση και χωρίς κράτος δικαίου δεν μπορούμε να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη. Αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Παρόλο που νέα κρούσματα σήμερα υπάρχουν μόνο στη Γουινέα, ε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θεώρησε τη Σιέρα Λεόνε και τις άλλες χώρες ζώνες ελεύθερες από τον ιό Εμπολά. Παρόλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες για να αποφύγουμε ε, νέα επιδημία σε περίπτωση αναζωπήρωσης ε, της, ε, των κρουσμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόιζερ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ησυχία των ΜΜΕ για την έμπολα είναι απατηλή. Υπάρχουν ακόμα κρούσματα στη Γουινέα και τη Σιέρα Λεόν και δεν είναι γνωστές ακόμα οι επιπτώσεις για τους επιζώντες της ε, ασθένειας. Είναι λοιπόν θετικό το ότι η έκθεση Γκέρνς μιλάει για πράγματα πέρα από την άμεση κατάσταση. Σημαντικό στοιχείο αυτό λοιπόν της έκθεσης αυτή Ευχαριστούμε Σάλς. Γι' αυτό παρακολουθούμε και ζητάμε την ενίσχυση των συστημάτων υγείας στις χώρες αυτές, Λιβερία, Γουινέα και Σχέρα Λεόνε, αλλά πρέπει να δούμε και τα άλλα ευπαθή και εύθραυστα κράτη της Αφρικής, όπως την κρίση των προσφύγων, όπου τα κράτη-μέλη με μισή καρδιά ασχολήθηκαν με τις αιτίε ε, της ε, κρίσης και εδώ πέρα υπάρχει μια έλλειψη γενικής ε, παροχής υγείας και υγειονομικών συνθήκων. Οπότε θα μάθουμε ότι το καλύτερο φάρμακο είναι η πρόληψη, ειδικά στην αναπτυξιακή συνεργασία. Φέτος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης πήγε δικαίως στο κουαρτέτο διαλόγου στην Ισία. Αυτό είναι θετικό. Οι άνδρες ε, και γυναίκες ε, οι οποίοι πήγαν να πολεμήσουν πρώτα απ' όλα την εμπολά ασθενείς και με νοσηλευτές και γιατροί και πολλοί από αυτούς πέθαναν επίσης θα άξιζαν το Νόμπελ Ειρήνης. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επιτροπή για τον ρόλο σας ως συντονιστής. Σας ευχαριστώ Γέρη και για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Στυλιανίδη, τι μαθαίνουμε μακροπρόθεσμα από την κρίση αυτή, πώς θα ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας των χωρών αυτών. Κύριε Γκέρνς, εγώ ασχολούμαι μια παρόμοια έκθεση για την ε, αντιπροσωπεία ΑΚΕ και μου λένε οι Αφρικανοί συνάδελφοι πως ε, εάν υπάρξει ξανά μια τέτοια πανδημία θα είμαστε εξίσου απροετοίμαστοι. Και ακούμε συνεχώς ε, ημωγές. Εγώ ζητάω να υπάρχουν παγκόσμια δίκτυα εκτάκτου ανάγκης. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες υποδομές για 24 ώρη ιατρική φροντίδα, αλλά θα πρέπει να σταματήσει και η διαφυγή των ιατρικών εγκεφάλων από τις χώρες αυτές. Χρειάζονται καλοί γιατροί εκεί πέρα και να τους εκπαιδεύσουμε. Και πρέπει να εμπλακούν και οι μητέρες στην υπόθεση αυτή αν ξέρουν και κάνουν το σωστό αυτό έχει χίλιες φορές μεγαλύτερη σημασία από το τι θα πει ένας Ευρωπαίος ε, που εργάζεται στην αναπτυξιακή συνεργασία. Ευχαριστώ. Σάντσες για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Γκέρνης, πρώτα πρώτα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους σας το επιτελείο για το άριστο έργο το οποίο επιτελέσατε σχετικά με την έκθεση από την κρίση του έμπολα που μας οδήγησε ε, τόσο θα να σας πω ότι η λιτότητα σκοτώνει και αυτό το οποία λέει το ΔΝΤ και η Διεθνή Τράπεζα και αυτό που κάνανε για τη δεκαετία του 80 επιδίνωσαν στην Αφρική ε, το σύστημα υγεία και οδηγήθηκαν σε αυτήν την κατάσταση με το έμπολο. Είχαμε περικοπές, είχαμε ιδιωτικοποιήσει ε, και στην Ευρώπη όπως έγινε στην Ισπανία και εκεί καταρρόξαν το, <clears throat> το σύστημα υγεία όπως είχαμε την Τερέσα Ρομέρο, την ε, νοσοκόμα, η οποία επειδή δεν υπήρχαν ε, όροι και μέσα, πέθανε. Επίσης τα ε, φάρμακα δόθηκαν μόνο για να κερδίσουν κάποιοι και όχι για να βοηθούν οι φτωχοί. Αυτό φάνηκε πιο πολλά. Είδαμε τι κάνει η λιτότητα για τα υγεία συστήματα υγείας, άρα θα πρέπει να βρεθεί κάποιο εναλλακτικό μοντέλο για την έρευνα για τα φάρμακα. Πρόκειται για κάποια παγκόσμια κρίση υγεία και για κατακλείδη να σα πω ότι αυτοί οι 12.000 νεκροί ε, θα πρέπει να το, μην επαναληφθούν. Χόιμπουχ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς οι πράσινοι ευχαριστούμε τον κύριο Γκέρεντς για την έκθεση και βεβαίως την χαιρετίζουμε γιατί πρέπει να λύσουμε διδάγματα για το μέλλον, για μελλοντικές κρίσεις γιατί αυτή δεν θα είναι η τελευταία. Τι θα θέλαμε εμείς σε αυτή την έκθεση. Θα θέλαμε να υπάρξει μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας γιατί εδώ πέρα αποδεικνύεται πως η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό. Γι' αυτό θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία δικαιωμάτων σε σχέση με τα φάρμακα. Και να προωθήσει το δικαίωμα των χωρών αυτών να εκμεταλλευτούν αυτά τα περιθώρια. Επίσης σωστή είναι η έκκληση που απευθύνεται σε όλες τις χώρες να υπάρχει μια σωστή και καθολική κάλυψη όσον αφορά τον προληπτικό τομέα της υγείας και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που υπάρχουν γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως ε, της κρίσης όταν περνάνε γιατί θα χρειαστούν πολλά χρόνια οι χώρες να τα ξεπεράσουν. Ευχαριστώ. Κυρία Γκίλ για ένα λεπτό. Α, ο κύριος Γκίλ με συγχωρείτε. Μάικ. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εξοπλίσω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τις τοπικούς συλλόγους που εργάζονται εντατικά κατά τη διάρκεια της κρίσης για το θάρρος που έχουν επιδείξει. Και είναι και ευκαιρία να ασκήσω κριτική τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για τον σκανδαλοθυρικό τρόπο με τον οποίο προέβαλαν αυτή την είδηση για να αυξήσουν τις μετρήσεις τηλεθέασης. Το BBC έχει Ebola Watch και αυτούς τους όρους τους χρησιμοποιούσε όταν ασχολιόταν με υποθέσεις εγκληματιών. Νομίζω ότι είναι τραγικό. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε όταν εξετάζουμε τις αιτίες και όχι τα συμπτώματα. Το πιστεύω ακραδάντως αυτό και μπορούν να προληφθούν ή να ε, μειωθούν οι τέτοιες κρίσεις με την αύξηση του πλούτου των πιο φτωχών στις πιο φτωχές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στερήσει από τους ανθρώπους της Δυτικής Αφρικής ε, τα προστοζήν και αυτό ε, ουσιαστικά ε, τους θέτει στο περιθώριο με την αλλιευτική της πολιτική βεβαίως. Έχουν χάσει την ευκαιρία να, να μπορούν να βρουν τα προστοζήν και να βελτιώσουν τις συνθήκες τις οποίες ζουν. Και γι' αυτό τέτοιου είδους κρίσεις θα συμβαίνουν ξανά και ξανά. Σαφχάουζερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Mes chers collègues. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμείς, ξέρετε, δεν, ε, δεν φοβόμαστε ε, το γελίο, γιατί το γελίο κυριαρχεί στην συνέλευσή μας απόψε. Έστω. Όμως, είμαστε γελίοι, γιατί ε, ξυπνάμε για τον έμπολα με 11.000 νεκρούς και αποδεσμεύουμε δυο δις, 900 εκατομμύρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της. Αλλά για την ελονοσία τι, 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν. 190 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί. 120.000 είναι αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη φροντίδα υγείας. Όμως υπάρχουν τα φάρμακα και δεν στοιχίζουν καθόλου αλλά αυτό δεν μας αφορά. Ε, νομίζω ότι έχουμε αποθρασυνθεί. Γιατί αυτό δεν μας αφορά και δεν φοβόμαστε ότι εμείς θα πληγούμε από την ελαιονοσία. Πότε θα έρθει το σχέδιο Μάρσαλ αυτό στην Ευρώπη. Έχουμε τρεις ε, ποσοτικής χαλάρωσης για τις τράπεζες. Έχουμε μια ψευδέστηση του Γιούνκερ υποτίθεται για την ανάπτυξη στην Ευρώπη και για την Αφρική τίποτα. Πανε Ebola zebrała największe żniwo w trzech krajach Afryki Zachodniej. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είδατε τι έγινε σε τρει ορθιδικέ από τον ε, ε, ιό αυτό σε Λιβερία, Γουινέα και Ρελιώνη. Οπότε αντέδρασε πάρα πολύ αργά η κοινότητα και επίση ε, και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Πέραν του ότι είδαμε τι τα συστηματικές αυτέ τι χώρε δεν υπήρχαν πόροι, δεν υπήρχαν δυνατότητε, ώστε να σταματήσει ε, αυτή η επιδημία ή οι επιδημίε αυτών όλων των ασθενειών αυτό ήταν ένα χτύπημα στην οικονομία όλης της περιοχής. Οι, δε, οι ε, οργανώσεις θα έπρεπε να βοηθήσουν τους ασθενείς και θα έπρεπε να τους προστατεύσουν. Όλοι αυτοί οι διεθνείς παίκτες να έχουν έναν ε, διάλογο, να έχουν συνεργασία με τις τοπικές αρχές και έτσι να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών που είχαν ε, πληγεί. Δεν θα έπρεπε να φοβάται ο κόσμος να ζητήσει βοήθεια και άρα θα έπρεπε να τους δοθεί ε, βοήθεια σε επίπεδο υγεία. Άρα θα πρέπει να εμπλακούν τα κράτη-μέλη σε κάποια πολιτική προπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Πρέπει να γίνουν επίση επενδύσει σε συστήματα υγεία. και έτσι θα φέρουμε οικονομική ανάπτυξη, θα καταβολήσουμε την ε, φτώχεια. Και επίση, στα πλαίσια του Horizon 2020 να βοηθήσουμε και με καινούργια φάρμακα. Να μισή λεπτό, κύριε Μάκρο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ και τον κύριο Γκέρενς και βεβαίως και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πέρα σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Έχετε δίκιο κύριε Επίτροπε. Το βασικό μάθημα είναι ότι εκεί που δεν υπήρχαν τα βασικά ενός συστήματος υγείας οι χώρες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Το ερώτημα μου είναι τι θα γίνει τώρα για να οικοδομήσουμε αυτά τα συστήματα υγείας έχει αλλάξει τίποτα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Τι θα γίνει στα κοινά μας προγράμματα με αυτές τις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Ε, φτιάχνουμε νέες κλινικές. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους εκεί. Με τις δεσμεύσεις που είχαμε στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο. Ε, και τα ρωτάω αυτά γιατί συνάντησα κάποιον που εργάζεται στη Σιέρα Λεόν σε Λεόνε και ε, έχει την εντύπωση ότι κάποιες εγκαταστάσεις διαλύονται, ότι δεν υπάρχουν γιατροί, ότι στη Σχέρα Λεόνε μόνο οι θυλάζουσες μητέρες και παιδιά κάτω των πέντε και οι έγκυες έχουν δωρεάν ε, παροχή υγείας. Ε, δεν υπάρχει τίποτα και για τους επιζώντες. Χρειάζεται ένα νέο πρόγραμμα υγείας και δεν ξέρω αν οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έχουν κάτι και αν συνεχίζουν να συντονίζουν. Γιατί όπως είπατε δεσμευτήκαμε στη Νέα Υόρκη για κάτι τέτοιο, αλλά δεν αρκεί η δέσμευση, πρέπει να το κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι λοιπόν σε αυτές τις χώρες. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια προς τον συνάδελφο Σαρλ Γέρνη για την έκθεση αυτή. Και τώρα όσον αφορά τα συμπεράσματα πρέπει να εξαγάγουμε για την ε, κρίση του ιού έμπολα. Πριν από μια εβδομάδα συνάντησα κάποιον εκπρόσωπο ενό μη κυβερνητικού από την Σιέρα Λεόνε. Πρόκειται για κάποια οργάνωση που καταρχήν ασχολείται με την παιδεία και μέσα στην κρίση του έμπολα ε, βρέθηκε εκεί στο επίκεντρο των προσπάθειων, ε, προσπάθειων για να σταματήσει η διάδοση της ασθένεια. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό ότι δηλαδή αυτή η κρίση ήταν κάτι σαν συναγερμό, σαν ξυπνητήρι και μας ε, έδειξε πού υπάρχουν όλα τα δύνατα σημεία των συστημάτων υγείας. Γιατί ήταν ανεπαρκής δηλαδή η αντίδραση. Οπότε θα πρέπει να υποστηρίξουμε, να αναβαθμίσουμε τα στήματα υγείας αυτών των χωρών και επομένως θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις σε σχέση με την χρηματοδότησή τους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και τώρα ξεκινούμε την διαδικασία. Διά, δεν θέλουμε ε, Και τώρα, η διαδικασία να ελκύσει στην προσοχή του Πρόεδρου. Κάτσε διά. Έχουν ε, εγγραφεί 10 ομιλητές. Όμως θα δώσουμε το λόγο σε έναν ομιλητή από κάθε πολιτική ομάδα, άρα έξι συνολικά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η επιδημία του 2014 ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία. Επηρέασε πολλές χώρες, πάνω από 20.000 άνθρωποι μολύνθηκαν, 5.000 πέθαναν. Πέθαναν επίσης και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έδωσαν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να αναπτυχθούν θεραπείες και εμβόλια. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει και παρέμβαση, ε, παρακολούθηση, ίχνη λάτηση, εκπαίδευση των ε, εργαζομένων στον κλάδο της υγείας και βεβαίως μια κοινωνική κινητοποίηση για να μειωθεί η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και βεβαίως ε, μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη περισσότερα για να βοηθήσει την ε, Δυτική Αφρική στη δοκιμασία που αντιμετωπίζει. Ευχαριστώ. Κινίτσι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μέγεθος και η δυσκολία αυτού του φαινομένου της ε, ασθενή χτύπησε Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα και οπότε έχει μεγάλη ευθύνη η Ευρώπη στην ε, διεθνή σκηνή ακριβώς γιατί θέλουμε να έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα υγείας και βοήθειας γιατί είδαμε ότι υπάρχουν διαρθρωτικέ ελλείψεις για την υγεία και εξαιτία των χτυπημάτων που δέχτηκαν αυτέ οι χώρε από την ασθένεια. Μα έδειξε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η κρίση. Οπότε και σήμερα ακόμα πιο επιτακτικό να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή βοήθεια και στην ε, υποστήριξη την οικονομική αυτών των τριών αφρικανικών χωρών. Και επίση συμφωνώ για όλα αυτά που λέει η έκθεση, όσον αφορά να έχουμε κάποια αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη και να βοηθήσουμε μέσω αυτού τι ε, τρει χώρε. Να έχουμε διαρθρωτική υποστήριξη και να βοηθήσουμε την προσβασιμότητα στην ε, υγεία και στις βασικές υπηρεσίε κοινωνικής προνοιάς ιδάλλως. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε και στο μέλλον τέτοια φαινόμενα επιδημία. Κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, από το 2014 η Σιέρα Λεόνε, η Γουινέα, και η λιβυρία πλήττονται από τον ιό του έμπολα ενώ άλλες πόλεις της αφρικής αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια κρούσματα του ιού. ωστόσο οι χώρες αυτές δεν βιώνουν μόνο την κρίση του ιού έμπολα αλλά γενικότερα μια συστημική κρίση αφού το 80% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. βέβαια η αντίδραση της ευρωπαϊκής ένωσης για περιορισμό του έμπολα δεν ήταν άμεση και ιδιαίτερα αποτελεσματική όπως ήταν οι γιατροί χωρίς σύνορα και ο ερυθρός σταυρός που αποδείχτηκαν περισσότερο προετοιμασμένοι για να βοηθήσουν τους πληθυσμούς της αφρικής για να αντιμετωπίσουν τον έμπολα. είναι επομένω αναγκαίο να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ικανότητες των ανθρωπιστικών αυτών οργανώσεων εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση να ενισχυθεί η ιατρική έρευνα για να παραχθούν φάρμακα και εμβόλια για τον έμπολα. επιπλέον είναι απαραίτητο να διαγραφεί το χρέο των χωρών τη Αφρική που έχουν πληγεί από τον ιό ώστε να μπορέσουν οι χώρες να επενδύσουν περισσότερα στα συστήματα υγείας τους αντί να πληρώνουν τους διεθνείς τοκογλύφους δανειστές διότι τα συστήματά τους αυτά έχουν διαλυθεί κυριολεκτικά από το διεθνές νομισματικό ταμείο. ευχαριστώ θα πρέπει να παίρνουμε κάποια μαθήματα από αυτή την κρίση του έμπολα. Οπότε για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να γνωρίσουμε τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ε, ακριβώς και έπληξαν τα συστήματα δημοσίας υγείας. Οπότε πάρα πολύ δύσκολο ήταν για αυτές τις χώρες να αντιμετωπίσουν αυτή την επιδημία. Θα πρέπει επομένως να σταματήσουμε αυτές τις ε, πολιτικές, να σταματήσει αυτού του είδους η υποδούλωση. Εμείς θέλουμε κάποιες παγκόσμιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Θέλουμε να υπάρχει κάποια κατάρτιση επαγγελματιών του κλάδου της υγείας. Να δούμε τι θα γίνει με τα διπλώματα βραστεχνίας ε, σχετικά με την φαρμακοβιομηχανία. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει εξυγίανση ε, των υποδομών, θα πρέπει να προσέξουμε ε, την πολιτική για την παροχή, γιατί είδατε τι έγινε με την Κούβα. Έστειλε πολύ περισσότερους ε, γιατρούς και ιατρικό προσωπικό από όσο όλες οι χώρες της Ευρώπης. Κύριε Ριβαζή. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ε, συγχαρώ τον συνάδελφο Γκέρενς για την ανάλυση του και για τις προτάσεις του. Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, άλλωστε μία από τις κόρες μου και ο γαμπρός μου εργάζονται στη Γουινέα, δύο κρούσματα έμπολα ξέσπασαν στο κέντρο ε, ε, του Ερυθρού Σταυρού στο Φουρεκαριά. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη έβαλαν στο τραπέζι πάνω από 1,9 δις ευρώ και τελικά δεν βελτίωσαν και τόσο τα συστήματα υγείας. Είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να γίνει. Ζητώ από τον Επίτροπο στο Ταμείο για την Ανάπτυξη να υπάρχουν εγγυήσεις ότι πράγματι με αυτά τα χρήματα θα φτιαχτούν νοσοκομεία και θα υπάρχουν τέτοιου είδους δυνατότητες. Από εκεί και πέρα δώσαμε κονδύλια για κλινικές μελέτες θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από αιρεσιμότητα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διπλώματα. Ε, ε, ε, Πατέντε κατοχυρωμένα για να μπορέσουν να γιατρευτούν οι άνθρωποι. Μία νοσηλεύτρια η οποία νοσηλεύθηκε ε, τελικά ε, υποτροπίασε και το σπέρμα περιέχει τον ιό έξι μήνες μετά τη θεραπεία υποτίθεται του ανθρώπου. Πρέπει να ξανα υπάρξει εμπιστοσύνη στα συστήματα υγείας από τους ανθρώπους που ζουν εκεί γιατί διακυβεύεται πραγματικά το μέλλον του. Ευχαριστώ. Οι γιατροί χωρίς ε, σύνορα, οι Σαμαρίτες, όλες οι ΜΚΟ κάναν καλή δουλειά. Ήταν εκεί επιτόπου να πολεμήσουν την αρρώστια πριν ξεκινήσουν και πριν το πάρουν καν χαμπάρι οι πολιτικοί. Και όταν κάναμε κάτι, κάναμε τα πάντα σε αργή κίνηση. Κυνηγούσαμε τα γεγονότα και για κάθε νέο νοσοκομείο που κάθε νέο νοσοκομείο που φτιάχναμε είχε γεμίσει μέσα σε λίγες ώρες. Αντί να επιτάξουμε υφιστάμενα δίκτυα, αρχίζαμε να, χτίζουμε, να χτίζουμε από το μηδέν και τα πράγματα χειροτέρευαν. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη και στις άλλες χώρες, την άλλη φορά αντιληφθείτε το κατεπήγον του πράγματος. Διδαχτείτε από τις ΜΚΟ, από τους ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους για να πολεμήσουν την έμπολα. Και ας μάθουμε το πάρα πολύ απλό, ότι το να δράουμε γρήγορα δεν είναι μόνο φτηνότερο, αλλά σώζει ζωές. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή την επικοδομητική και τις προτάσεις σας. Θα ήθελα να επαναλάβω πως η έκθεση Γκέρενς μας δίνει κάποια πολύτιμα μαθήματα. Όλοι αντλούμε διδάγματα από αυτή την υπόθεση ακόμη μια φορά. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τσάλς Γκέρενς για τη δουλειά που έκανε. ταυτόχρονα. Θα ήθελα να πω κάτι για αυτό το οποίο είπε η κυρία Μακάμαν για ένα σύστημα καθολικής παροχής υγείας. Όπως είπα ήδη συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό ακριβώς και συζήτησα και εστίασα στο πρόβλημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει μεγάλη σημασία το θέμα αυτό για την επόμενη εκδήλωση της ασθένειας. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προωθήσουμε το ζήτημα αυτό για να προλάβουμε την επόμενη επιδημία. Βεβαίως, Κομισιόν και κράτη-μέλη πρέπει από κοινού να ξαναδούνε την αναπτυξιακή συνεργασία στον τομέα της υγείας, ειδικά στις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Είδα επιτόπου εγώ τα προβλήματα των τριών χωρών και συνειδητοποίησα ότι τα μαθήματα που αντλούμε είναι η σημαντικότερη βάση για το μέλλον, για εμάς, την διεθνή κοινότητα και βεβαίως πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις χώρες ε, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και βεβαίως ε, πρέπει να δούμε τους στόχους της χιλιετίας που έχουν σχέση με την υγεία και βεβαίως να έχουμε ανθεκτικά συστήματα υγείας για να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για τις μελλοντικές εκδηλώσεις της ασθένειας. Γιατί θα έχουμε ξανά βεβαίω κρούσματα. Πρέπει να γίνει αυτό με τρόπο πιο στοχευμένο και προβλέψιμο μακροπρόθεσμα μόνο έτσι γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Γκέρνς για την ε, δουλειά που έκανε. Γιατί τώρα έχουμε μια βάση για τις ε, μελλοντικέ μας ενέργειες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Γκέρντς. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς θα ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στο πλαίσιο συζήτησης της έκθεσής μου. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για το άτομό μου. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Στυλιανίδη για τη συνεργασία. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά, επίκαιρα, είναι θέματα ζωής και θανάτου και πρέπει να τα πάρουμε πολύ σοβαρά. Η Επιτροπή μας για την Ανάπτυξη ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες εδώ και χρόνια επιμένει στην ανάγκη να δοθούν περισσότερα μέσα στην προώθηση του κλάδου της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Επιτροπή μας αξιοποίησε κάθε δυνατή ευκαιρία και στις συζητήσεις για τον προπολογισμό και στις συζητήσεις για ειδικέ εκθέσεις για το θέμα αυτό ε, επέμεινε σε κάθε ευκαιρία να δοθούν περισσότερες δυνατότητες έρευνας στις αφρικανικές χώρες, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα στις αφρικανικές χώρες. Δεν αναπτύσσουμε τους άλλους. Πρέπει να δώσουμε στους άλλους μέσα και εργαλεία να αναπτυχθούν μόνοι τους. Και σε κάθε ευκαιρία επιμείναμε στη βελτίωση της διακυβέρνησης σε παγκόσμιο, διεθνές, ευρωπαϊκό ή αφρικανικό επίπεδο. Δεν υπάρχει τίποτα το πεπρωμένο θα έλεγα ε, και μοιραίο γιατί είχαμε αποτελέσματα. Ε, σε όλες τις ευκαιρίες ε, επικρίναμε την βραδύτητα των αντιδράσεων της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών φορέων και οργανισμών και τελικά δρομολογήθηκαν τα πράγματα. Και κυρίως χάρη στο ψήφισμα το οποίο ψηφίσαμε το Σεπτέμβριο του 2014, το οποίο ήταν κατά την άποψή μου το καλύτερο ψήφισμα που έχουμε εγκρίνει ποτέ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που να αφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είπε κάποιος συνάδελφος ότι είμαστε γελοί και έκανε την αντιπαραβολή μεταξύ ελονοσίας και έμπολα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν λέμε ή το ένα ή το άλλο. Εμείς λέμε και το ένα και το άλλο. Και τον έμπολα πρέπει να πολεμήσουμε και την ελαιονοσία. Δεν ε, διαλέγει κανείς να πολεμήσει ή τη φυματίωση ή το AIDS και τα δύο ε, ε, προσπαθεί να πολεμήσει και αγωνίζεται να λύσει αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να αυξηθεί η ενίσχυση που δίδεται κατά 20%. Εμείς όμως αυτό το έχουμε ε, εγκρίνει και μας λέει γελίους και ήρθε εδώ για να μας πει γελίους και να φύγει ένα λεπτό αμέσω μετά. Δεν θα πρέπει να ε, σταματήσουμε να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι ένας ιός τρομακτικός, ο οποίος μεταλλάσσεται, προκύπτει ξανά και ξανά, με διαφορετικές μορφές, με διαφορετικές οδούς μετάδοσης. Δεν έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ακόμα. Πρέπει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί. Και τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει θα μας βοηθήσουν και πιστεύω ότι στα τέλη του 2015 είμαστε σε τελείως διαφορετική ε, κατάσταση συγκριτικά με το, την περίοδο κατά την οποία ξέσπασε η κρίση του αέμπολα το 2014 το φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο μήνυμα να στείλω. Η έκθεση επιμένει επίσης στο θέμα του ποιος είναι υπεύθυνος για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Η αγορά έχει σημαντικό ρόλο να παίξει, αλλά δεν θα πρέπει να την αφήσουμε μόνη της. Και εγώ, ξέρετε, είμαι υπέρ της ανάπτυξης της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Ωστόσο υπάρχουν ολόκληροι τομεί στην οικονομία που οι πολιτικοί θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και ελπίζω ότι το περιβάλλον, η η υγεία, οι αντίστοιχες κοινοβουλευτικέ επιτροπές περιβάλλοντος υγείας και βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα συνεργαστούν για να βρεθούν ακόμα καλύτερες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα το οποίο είναι εξαιρετικά ακαθόδε Και μάλιστα ε, γι' αυτό δεν το περιλάβαμε το θέμα αυτό το συγκεκριμένο στην έκθεση ε, τόσο εμπεριστατωμένα και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τα λεγόμενά μας και να ασχοληθεί περισσότερο σε βάθος με αυτό το εξαιρετικά ε, σημαντικό σημείο. Ευχαριστώ.